Καλημέρα σας. Ε, συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας σήμερα με τον πρέσβη κύριο Τότ που είναι ο υπεύθυνο ε, για ο εκτελεστικό γραμματέα τη οργάνωσης για τη συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών που είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ και είναι πολύ επίκαιρο αυτή την εποχή. Είστε εκτελεστικό γραμματέα αυτής της οργάνωσης ε, ήδη κάμποσο καιρό. Έχετε μεγάλη πείρα όσον αφορά τον αφοπλισμό και η συνθήκη αυτή τη πλήρου απαγόρευση. Ε, πρέπει να προσυπογραφεί υπογραφεί από 44 κράτη ε, για να ισχύσει και ακόμη ελείπονται 9. Οπότε θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την κύρωση αυτή και όσον αφορά την επικαιρότητα της περασμένης εβδομάδας, γιατί ήσασταν και εσείς στη Νέα Υόρκη για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ήταν ε, αφιερωμένο στην ε, ε, μη εξέλιξη ε, κύριε Πρέσβη, σας δίδω το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία διότι νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα, για την οργάνωση, να εκφράσω την, ε, ε, την ε, ευγνωμοσύνη μου για την συνεχή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις προσπάθειές μας και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, όπως άλλωστε το είπε ο κύριος Νοζό, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα ε, η οποία πέρασε σε επίπεδο προέδρων και πρωθυπουργών για την ε, ε, μη επέκταση των πυρνικών δοκιμών και τον αφοπλισμό. Θα αναφερθώ στην πρόοδο της συνθήκης και της οργανώσεώς μας τα τελευταία χρόνια παρόλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε ακόμη και θα ήθελα να αναφερθώ ε, και ε, στην όθηση ε, που έχουν οι προσπάθειές μας και θέλω να σας εξηγήσω γιατί χρειάζεται η συνθήκη αυτή και ο μηχανισμός επαλήθευσης. Ξεκινώ με πρώτα στοιχεία και ορισμένες πληροφορίες η ε, η συνθήκη αυτή ανέρχεται στο 1996 που υπογράφηκε για πρώτη φορά και απαγορεύει ε, τις πυρηνικές ε, ε, δοκιμές, δοκιμές πυρηνικών όπλων για πάντα. Είναι ένας συνδυασμός συνθήκης απαγόρευσης που συνδυάζεται με ένα καθεστώς επαλήθευσης και τα δύο συστήματα συνυπάρχουν. Ο ο κύριος Ντονζό με πρόλαβε ε, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε που είναι μοναδικός διότι ε, υπάρχουν 44 χώρες οι οποίες καθορίζονται στη συνθήκη και για να ισχύσει η συνθήκη πρέπει να έχουν κυρώσει και οι 44. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δικηγόρων τουλάχιστον που επενόησαν ένα τέτοιο σύστημα και ελπίζω ότι είναι και η τελευταία φορά. Είναι λοιπόν ε, ε, διπλή η χαρά για μένα. Όσον αφορά την πρόοδο και εδώ σε περίπτωση που έχετε ανοίξει τον προβολέα ίσως χρειάζεται λίγος χρόνος θα μπορούσε ο συνάδελφός μου να σας δείξει ορισμένες διαφάνειες αλλά προς το παρόν θα προσπαθήσω να χρωματίσω την ομιλία μου με τις διαφάνειες το σύστημα επαλήθευσης εξασφαλίζει ότι η απαγόρευση εφαρμόζεται και αποτελείται από τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ένα συνολικό σύστημα παρακολούθησης το οποίο ακούει ελπίζουμε ε, την ε, ε, σιωπή ε, των δοκιμών, την απουσία δηλαδή στην ατμόσφαιρα ήχων σχετικά με τα πυρηνικές δοκιμών ή στο, στην ατμόσφαιρα, στη γη, στη θάλασσα, στους ωκεανούς και αν υπάρξει οποιοδήποτε ήχος έχουμε πάνω από 300 ε, ε, οργανώσεις. Έχουμε δηλαδή καλωδιώσει ολόκληρο τον κόσμο. Ακούμε τα, ε, το τι γίνεται και υπάρχει τεχνολογία η οποία θα εντοπίσει αμέσως την ύπαρξη μίας έκρηξης. Όλες ε, αυτές, ε, όλοι αυτοί οι ήχοι που συγκεντρώνει και η τεχνολογία λοιπόν αποστέλλονται στον εγκέφαλο, στη Βιέννη, στο Διεθνές Κέντρο ε, Συλλογής στοιχείων όπου ε, υπάρχει ε, το κέντρο που συνδυάζει 250 εγκαταστάσεις επικοινωνίας ανά τον κόσμο. Θα σας δείξω μετά ένα, μία διαφάνεια διότι υπάρχουν πολλοί ήχοι βέβαια. Στη Σαμόα εχθές ακούσατε ε, ότι είχαμε ένα σεισμό 8 ρίχτερ συν τσουνάμι. Οπότε οι εγκαταστάσεις αντιλαμβάνονται και καταγράφουν αυτούς τους ήχους αλλά δεν μας ενδιαφέρουν για την παρακολούθησή μας και πρέπει να διαφοροποιήσουμε το τσουνάμι, τον σεισμό και ε, κάτι το οποίο είναι ανεξήγητο δια των φυσικών ε, ε, γεγονότων και αυτό κάνουμε στη Βιέννη. Άπαξ λοιπόν και συλλεγούν οι πληροφορίες δεν, ε, δεν είμαστε μία παρκετέζα που απλούστατα αφομοιώνει και ρουφάει τη σκόνη και την αδειάζουμε κάθε δύο χρόνια παραδείγματο χάρη αλλά ε, είναι ένα κέντρο επαλήθευσης των πληροφοριών και μόλις έχουμε τις πληροφορίες τις αντικατοπτρίζουμε στο σύστημά μας ε, σε 1200 χρήστες σε πάρα πολλές χώρες και γι' αυτό θα σας εξηγήσω μετά δεν, ε, γιατί με μεταφέρονται όλα αυτά τα gigabytes ε, στοιχείων ανά τον κόσμο. Πρόκειται για ένα ε, σύστημα που ονομάζεται, είναι το δίχτυμα ασφαλείας, δηλαδή είναι ε, το τρόπος παρακολουθήσεως και ε, γίνονται κατόπιν αυτού επιτόπιες ε, επιθεωρήσεις εάν δηλαδή ε, κάποιος θεωρηθεί ότι έχει προβεί σε μία έκρηξη αμέσως πηγαίνουμε επιτόπου με πολύ εξελιγμένη τεχνολογία να παρακολουθήσουμε τι έχει γίνει και τον παρακολουθούμε και πολύ πιο στενά για το επόμενο επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα το σύστημα αυτό ισχύει από το 1997 όταν άρχισε να λειτουργεί ο οργανισμός αυτό στη Βιέννη. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σύστημα το οποίο βλέπετε στο χάρτη πρόκειται για 600 διαφορετικές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο, πραγματικά σε όλο τον κόσμο, διότι έχουμε ε, σταθμούς στην Ανταρκτική, σε απόμακρα νησιά που δεν υπάρχει καν σύνδεση με με πλοίο τακτική και άλλες εγκαταστάσεις είναι σε, ε, ε, σε διοικητικά κέντρα. Πρόκειται για εγκαταστάσεις κόστους ε, πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχει προσωπικό το οποίο λειτουργεί το σύστημα από τη Βιέννη και έχουμε και περίπου 700 άτομα που απασχολούνται στα διάφορα κέντρα με τον κόσμο. Ε, το, το, πρώτο, το, πρώτο σύστημα απετέλεσε το πρότυπο και ε, έχουμε τώρα αρκετές εγκαταστάσεις το σύστημα αυτό δυστυχώς δοκιμάστηκε δύο φορές και ε, διαπιστώθηκε ότι η Κορέα το 2006 και το 2009 έκανε δύο πυρηνικές δοκιμές και θα δείτε ίσως ή στη διαφάνεια πως οι διάφοροι σταθμοί ανά τον κόσμο ενετόπισαν το σεισμικό σήμα μιλάμε ε, για ε, πολλούς ε, σταθμούς και το πολιτικό μήνυμα διπλωματικά για τα 61 συστήματα τα οποία παρακολουθούσαν θυμάστε ότι στο Ιράκ η πηγή της επαλήθευσης των πληροφοριών το γεγονός του εάν ε, η ε, πληροφορία προέρχεται από μία ή από περισσότερες πηγές πώς μπορεί κανείς ε, να χαλκιδεύσει τα στοιχεία εδώ εδώ προσπαθούμε να μην μπορεί κανείς να επέμβει στα στοιχεία αυτά στο μέτρο του δυνατού και να υπάρξει μία ουδέτερη επαλήθευση των στοιχείων μέσω των πολλαπλών συμφωνιών και οργανώσεων ε, που συμμετέχουν ή στην πλήρη απαγόρευση. Εκτός των σεισμικών συστατικών που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της 25ης ε, Μαΐου. Ε, θα σας δώσω ε, ένα παράδειγμα από την πρώτη ποινική δοκιμή της Βορείας Κορέας όπου η έκκληση 2,5 κιλοτόνων ενός αερίου το οποίο διαχύθηκε πρόκειται για ένα μπλε αέριο το οποίο ε, εκλείεται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αλλά έφτασε στην Νότιο Ασία μετά από κάποιο χρόνο. Βλέπετε λοιπόν ότι το σύστημα ε, είναι αποτελεσματικό. Ε, η έκρηξη που ήταν πολύ πιο μικρή από αυτές άλλων χωρών μπορεί να εντοπιστεί μέσω της εκκλήσεως αυτού του αερίου και έχουμε τώρα το σύστημα αυτό σε λειτουργία και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα πιο κοντινά συστήματα προς το σημείο της εκκλήσεως. Πρόκειται λοιπόν για ένα μηχανισμό προτύπου παρακολουθήσεως ε, της, ε, της εκρήξεως και ε, υπάρχουν 30 διαφορετικές πλατφόρμες ορισμένες σε πλοία, ορισμένες σε αεροπλάνα, άλλες στη γη είναι ε, το είδος των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τις μετεωρολογικές προβλέψεις και ε, βλέπετε ότι βασιστήκαμε, είχαμε βασιστεί σε προσωμιάσεις από τα στοιχεία που συνέλεγαν ε, οι 600 σταθμοί ανά τον κόσμο ε, για να εντοπίσουμε και την έκρηξη στην Κορέα. Το πιο βασικό λοιπόν εδώ είναι να επιτρέψουμε στις χώρες να εξασφαλίσουν ότι καταρχήν θα υπάρξει μία απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών για όλους που θα γίνει σεβαστή από όλους και να γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει. Δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικό αρνητικό ή θετικό σήμα σε, στην απαγόρευση των πυρνικών δοκιμών διότι ε, θυμάστε ότι τα τελευταία χρόνια οι πορισμένες περιπτώσεις ε, μπορεί και η αρνητική και η θετική δύναμη να αποτελέσουν προβλήματα και ε, ε, ε διαπιστώσαμε ότι από το 2000 ε, μέχρι τώρα 250.000 περιπτώσεις εκ των οποίων δύο ήταν μόνο σχετικές με την συνθήκη, δύο πυρνικές κρίξεις δηλαδή και πρέπει να πω ότι είναι δύο βελόνες σε μία θυμονιά 250.000 περιπτώσεων πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι δεν ε, έχει παρερμηνευθεί ε, η φύση των ε, άλλων κρίξεων και στην οργάνωση αυτή συμμετέχουν πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών έχουμε μία ενδιαφέρουσα κατάσταση διότι ξέρετε ότι στα τελευταία 8-9 χρόνια οι Ηνωμένε Πολιτείες Ε, είχε, είχε ε, ορισμένους ενδιασμούς για τη συνθήκη αυτή αν θα έπρεπε να είναι πολύ δεσμευτικό και τα τελευταία ε, εννέα χρόνια παρόλα αυτά οι Ηνωμένε Πολιτείες στο σύνολο του ενός δισεκατομμυρίου επένδυσης κάλυψαν τα 200 εκατομμύρια και από τις 42 ε, ε, ε, εγκαταστάσεις τις οποίες αποσκοπούμε ισχύουν ήδη οι 39 πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο την δυνατότητα να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία αλλά και να υπάρξει πολυμερή συνεργασία για να υπάρξουν ανταλλαγές πληροφοριών. Βλέπετε λοιπόν ότι ότι ακόμη και η πιο προηγμένη τεχνικά χώρα ενδιαφέρεται για το σύστημα αυτό ενώ στην αρχή δεν ήταν τόσο ενθουσιώδης για την επαλήθευση από πολυμερείς οργανισμούς το θέμα είναι ότι θα πρέπει κανείς να μπορεί να λειτουργήσει και να διαχειριστεί ένα τέτοιο σύστημα το οποίο είναι επιστημονικά πολύ πολύπλοκο όπως είναι αυτό το οποίο χρειάζεται 10.000 ε, χρόνια επιστήμης για να μπορέσει να λειτουργήσει. Λοιπόν, ε, καταλαβαίνετε ότι μέχρι το 2009 είστε από την Κοσταρίκα που δεν έχει καν στρατό επισήμως ε, αλλά που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας για να εξετάσει κάποια δοκιμή. Είναι ε, διαφορετικό από το να, ξέρετε τι έχει συμβεί προηγουμένως ή να πρέπει κι εσείς να συζητήσετε ισότιμα με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με το σύστημα λοιπόν αυτό μια μισή ώρα ε, ε, με από την έκρηξη 112 ε, πρωτεύουσες ε, γνώριζαν ε, το, την έκταση της έκρηξης διότι υπήρξε μια σεισμική δόνηση 5 χιλιόμετρα από εκεί που είχε γίνει η προηγούμενη πυρνική δοκιμή. Τέτοια πράγματα δεν είναι συνηθισμένα εάν εάν είναι βαθιά μέσα στη γη ενδέχεται να είναι σεισμός. Αν είναι όμως στην επιφάνεια τότε είναι κάτι ε, κάτι διαφορετικό. Σε νέα λοιπόν το πρωί στις 25 Πέμπτου 2009 συγκαλέσαμε τους ενδιαφερομένους, τους δείξαμε ποια είναι ε, τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, τη διαφορά από το σεισμογράφο ε, ενός σεισμού και το σεισμογράφο και το αποτύπωμα αυτού του γεγονότος και η Αυστρία, η Κωνσταντίνα, η Μπουρκίνα Φάσο, η Τουρκία, το Βιετνάμ, η Ουγγάντα ε, ισότεμα γνώριζαν τι είχε συμβεί. Βέβαια όλοι αυτοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν πολιτικά στο ίδιο επίπεδο αλλά η κρίση τους βασίζεται σε στοιχεία τα οποία αποτελούν σαφείς πληροφορίες από μία ε, πηγή η οποία στηρίζεται από πολλές χώρες οι οποίες, όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις αυτές. Υπάρχει λοιπόν μία ισότιμη αντιμετώπιση και το σύστημα αυτό όπως βλέπετε δυστυχώς απεδείχθη ε, επιτυχές μπορεί όμως να χρειαστεί και στο μέλλον αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι το σύστημα αυτό είναι μοναδικό. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι και οι απαγορεύσεις είναι μοναδικές διότι για πρώτη φορά στην ιστορία της, του αφοπλισμού και της απαγορεύσεως των πυρνικών όπλων οι διάφορες χώρες δεσμεύουν και τους οπλισμούς τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η σημασία αν γνωρίζετε τις λεπτομέρειες αυτών των συνθήκων. Λοιπόν είναι ένα περιβάλλον το οποίο θα ισχύσει για πάντα και θα επηρεάσει τους πάντες. Το άλλο βασικό είναι ότι οι υποχρεώσεις επαλήθευσης είναι οι ίδιες. Υπάρχει μία υποχρέωση η οποία έχει αναλυφθεί για πρώτη φορά να εκτίθενται ε, οι ενδιαφερόμενοι σε επαληθεύσεις ε, ανα πάσα στιγμή, πράγμα το οποίο έχει επίσης σημασία Οπότε ένα τρίτο των σταθμών που είδατε στην πρώτη διαφάνεια βρίσκονται από, από τα 340, από 340 σταθμούς οι 110 είναι στις χώρες που έχουν πυρηνικούς οπλισμούς και αυτές ε, συμβάλλουν ε, διότι υπήρχαν ε, προηγούμενη σταθμή σταθμοί ε, πυρηνικών ε, δοκιμών εκεί και καμία χώρα ακόμη και η μεγαλύτερη δεν θα μπορούσε να κατασκευάσει ή να λειτουργήσει αυτές τις εγκαταστάσεις μόνης της η κατανομή των στοιχείων είναι δημοκρατική όπως σας είπα ο τρόπος μετάδοσης των πληροφοριών είναι μοναδικός και μπορούν όλες οι χώρες να αισθάνονται ενήλικες και ισότιμες στην, στη διεθνή κοινωνία. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση της ενάρξωσης χείρος διότι από τα 44 ονόματα όπως σας είπα 9 ακόμη υπολείπονται ε, όσο ε, ε, το Πακιστάν, η Ινδία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Ινδονησία μας προβληματίζουν αλλά το ευχάριστο είναι ότι από το 1997 από μηδέν κυρώσεις έχουμε φτάσει σε ένα σύνολο 150 και 35 από τις 44. Ε, αν λοιπόν ε, αν λοιπόν σκεφτούμε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια δεν ήταν η χρυσή εποχή των πολυμερών σχέσεων ε, και σκεφτείτε ότι κυρώθηκε η συνθήκη αυτή από 100 επιπλέον μέλη ε, πιστεύω ότι υπάρχει πεποίθηση ε, πεισματικά στην διεθνή κοινότητα ότι πρέπει να ισχύσει αυτή η συνθήκη και ότι το σύστημα αυτό επαλήθευσης είναι χρήσιμο. Διαφορετικά δεν πρόκειτο να κυρώσουν 100 κράτη εν λευκό και ε, ε, πολλές φορές γνωρίζουν ότι μέσω αυτής της κυρώσεως ενοχλούν στρατηγικούς εταίρους και επίσης ε, υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες δεν θα μπορέσουν να υλοποιήσουν ορισμένα προγράμματα κατά αυτόν τον τρόπο τα γεγονότα της, τελευταίας εβδομάδος μας ε, επιβεβαίωσαν ε, διότι την περασμένη εβδομάδα κατόπιν προσκλήσεως του Πρόεδρου Ομπάμα ε, ε, ε, υπερψηφίστηκε το ψήφισμα 80-87 για, την, για να ισχύσει η συνθήκη για την απαγόρευση πυρηνικών δοκιμών πιο νωρίς μόνο ο, τρεις τέτοιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν υπάρξει στα τελευταία 16 χρόνια και ε, θυμάστε ότι η συνθήκη αυτή υπογράφτηκε το 1996 Άρα αυτό είναι μία σαφής ένδειξη για οποιονδήποτε το αμφισβητεί ότι τουλάχιστον όσον αφορά το μυαλό του Προέδρου ο στόχος αυτός ισχύει. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το στόχο αυτό και εδώ η συνδρομή σας και όλων αυτών που πιστεύουν στους κανόνες δικαίου σε πολυμερίες περιβάλλον σε εξίσου με, με εξίσου δεσμευτικό τρόπο ε, θα μπορέσουν να συμβάλλουν στο να εφαρμοστεί η ιδέα αυτή. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει στις ανατολικές χώρες, τι θα γίνει στην Ινδία, στο Πακιστάν, στο Ισραήλ, στο Ιράν και στην Αίγυπτο. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά αν ε, ενδιαφέρεστε, ε, στη δεύτερη φάση. Η συνθήκη αυτή όμως είναι ένα απαραίτητο τμήμα του καθεστώτος ε, πλήρους απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών και βλέπουμε ότι Υπάρχει, ε, ε, υπάρχουν ορισμένες ατέλειες στο καθεστώς αυτός και ε, του χρόνου θα γίνει μία συνεδρίαση διότι θα πρέπει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι στη διάθεση όλων δηλαδή όλοι να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα διότι δεν δούμε μόνο σε ένα περιβάλλον μετά την 11η Σεπτεμβρίου αλλά και μετά την επίθεση στο Μουμπάι, στο Ισλαμαμπάντ σε ένα περιβάλλον όπου η κατάχρηση των ε, δυνητικών ε, ε, πυρηνικών υλικών ή σχάσιμων υλικών αποτελούν κίνδυνο για όλους μας. Οπότε ε, χωρίς αυτή τη συνθήκη το καθεστώς αυτό θα μπορέσει ίσως να επιβιώσει μερικά χρόνια ακόμη αλλά δεν θα είναι βιώσιμο ε, για μεγαλύτερη διάρκεια γιατί είναι η τελευταία γραμμή αμήνης η συνθήκη αυτή. Αν η Βόρειος Κορία ακολουθήσει τον λάθος δρόμο θα χρειαστεί να περάσει αυτό το τελευταίο εμπόδιο. Αν λοιπόν ρωτάτε για ποιο ε, είναι ε, ε, το προσόν αυτής της συνθήκης έναντι μία τόσο πείσμονος χώρας, υπάρχουν οι δυνατότητες να κινητοποιήσει κανείς τη διεθνή κοινότητα. Πρώτα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επίπεδο που δεν γίνεται σεβαστό και μετά θα δούμε ότι η ε, διεθνής κοινότητα έχει τη δύναμη τη, η οποία βασίζεται σε αποφάσεις του Βουλίου Ασφαλείας. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ και μετά θα σας δώσω τις απαντήσεις αν το επιθυμείτε. Ευχαριστούμε για αυτές τις τεχνικές επεξηγήσεις που ήταν σαφείς και πολύ χρήσιμες. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Λούζινγκ πρώτη και καλύτερη. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για αυτή την λεπρομενή και πολύ επιγγερματική παρουσίαση του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε μόνο να χαιρετήσουμε. Χαιρετίζω επίσης και το ψήφισμα το, στο οποίο αναφερθήκατε διότι αυτό το ψήφισμα όντως μας οδηγεί ε, να ε, πιστεύουμε ότι αυτή η, ε, η διαδικασία που καθυστερεί όντως αποτελεί, αποκτά μια νέα δυναμική. Αναρωτιέται κανείς πώς αυτές οι χώρες δεν ε, κυρώνουν αυτές, αυτή τη συνθήκη. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις ή διαφορετικά συστήματα ε, όσον αφορά την πολυπτυχή πτυχή και την στρατιωτική πτυχή ε, διότι ο πρόεδρος Ομπάμα ζητά να κυρωθεί ο ίδιες όμως οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν κυρώσει. Άρα θα θέλαμε να ξέρουμε ε, πώς μπορεί κανείς να, έχει πει, να εξασκήσει πίεση στις Ηνωμένε Πολιτείε στο Ισραήλ. Ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι υπάρχουν και για συγκεκριμένους τεχνικούς ή στρατιωτικούς λόγους δεν προβαίνουν στην κύρωση Ίσως είναι τεχνικά θέματα τα οποία αναφέρω σχηματικά, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι η στρατιωτική ε, κύκλη στις Ηνωμένε Πολιτείες πολλές φορές ε, αναφέρονται στην δυνητική χρησιμοποίηση ε, πυρνικών όπλων όπως ο Ρόμπερτ Χούπερ. Το πιο πιθανό σενάριο το οποίο τον έχω διαβάσει είναι ότι ε, μπορεί αυτό να γίνει ε, για να καταστραφούν ε, κρυμμένα βιολογικά όπλα είναι όμως πυρηνικά όπλα τα οποία δεν μπορούν να εξελιχθούν χωρίς, ε, χωρίς δοκιμές. Άρα εσείς θεωρείτε ότι ενδέχεται η στρατιωτική κύκλη των Ηνωμένων πολιτιών ε, σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Πρόεδρου Ομπάμα να θελήσουν ε, να μην κυρώσουν για αυτούς τους λόγους. Ο κύριος ε, ε, Σφόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα πριν από λίγο καιρό τη δυνατότητα ε, επειδή το γραφείο αυτό δεν είναι πολύ μακριά από το σπίτι μου να τους επισκεφθώ και ήθελα και τους έκανα ορισμένους, ορισμένες ερωτήσεις αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο έχει επαφές με τις Ηνωμένε Πολιτείε, επισκέπτεται τις Ηνωμένε Πολιτείε όπου υπάρχει επίσημη ε, αμερικανική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία και εις ε, τις διασκέψεις κορυφής ε, διατυπών εκδηλώνει ψήφισμα το Κοινοβούλιο θα πρέπει ίσως να στηρίξουμε αυτά τα οποία μας είπε ο πρέσβης δηλαδή ε, πρέπει να δούμε πως ε, χωρίς ε, να το λάβει υπόψη της η δημόσια γνώμη έχει καταρτιστεί ένα πολύ ενδιαφέρον και καλό σύστημα επαληθεύσεως και άρα διακομματικά μέσω των επαφών μας με τους γερουσιαστές ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε θα έπρεπε να εκδηλώσουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κίνηση αυτή διότι αν κυρώσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πιέσουν και τις άλλες χώρες δεν μπορεί να πιέσει δεν μπορεί να πιέσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε μία χώρα άλλη να υπογράψει εφόσον αυτή αυτοί δεν το έχουν πράξει. Ευχαριστώ. Κύριος Βάιγκελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που αναλάβατε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιες οργανώσεις συνδέονται με το βασικό θέμα της υποεπιτροπής μας. Καμιά φορά όμως είναι δύσκολο να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μας και για τις πρόσφατες εξελίξεις. Και εγώ είχα παρόμοια θέση στη Βιέννη πριν από πολλά χρόνια και 10 χρόνια και χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος. Όταν ήμουν στη Βιέννη όλα αυτά ήταν στα χαρτιά ακόμη, ενώ τώρα βλέπω ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλά, πολλές από εκείνες τις ιδέες. Το κύριο λοιπόν πρόβλημα το έθιξαν οι συνάδελφοι και υπάρχει ακόμη ότι ορισμένες χώρες είναι ακόμη, ε, αρνούνται ακόμη να συμμετάσχουν και αυτό δημιουργεί όχι μόνο προβλήματα διάδοσης αλλά όντως πραγματικών σειράξεων και άλλων κινδύνων που αντιμετωπίζουμε παγκόσμια. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία λοιπόν να καταφέρουμε το Ισραήλ ας πούμε να συνδεθεί με αυτήν τη συνθήκη ή την Κίνα ή το Ιράν, το Πακιστάν. Δέχομαι βέβαια με ικανοποίηση το γεγονός ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν πάρει πια μια πιο επικοδομητική θέση και ελπίζω και η συζήτησή μας να συμβάλλει στην καλύτερη γνωστοποίηση των θεμάτων αυτών και από την κοινή γνώμη και από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι φανερό ότι και όπως είπατε και εσείς οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εδώ το προβάδισμα. Εσείς βέβαια ως διπλωμάτης δεν μπορείτε να τα πείτε όλα καθαρά, αλλά είναι φανερό ότι τα στοιχεία είναι ένα πράγμα και η χρησιμοποίησή τους άλλο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ξέρω πώς μπορούν να παρέμβουν στη Σλοβενία ή την ακτή του Ελεφαντοστού. Καλό είναι λοιπόν οι δεσμεύσει και υποσχέσεις να συμβαδίζουν, να συνοδεύονται από πραγματική διάθεση πραγματοποίησης των κοινών μας στόχων. Δεν είδα όμως στην πληροφόρησή σας κύριε Πρεσβευτά να λέτε τίποτε για περισσότερη προθυμία της Ρωσίας για συνεργασία. Ίσως μπορείτε να μας πείτε κάτι και γι' αυτό. Τι συμβαίνει με τη Ρωσία, με τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Ένα αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ για την ε, τόσο κατατοπιστική τοποθέτηση. Και εγώ, όπως οι προλαλήσαντες, πιστεύω ότι το επίκεντρο αυτής της νέας ελπίδας που προδιαγράφεται μέσα στη συνθήκη του CPBT είναι η θέση των ΙΠΑ και θέλω περισσότερες ε, πληροφορίες ε, για το τι ε, συμβαίνει στην ε, Γερουσία, ποιες είναι οι συζητήσεις. Η Γερουσία χθε αντέδρασε αρνητικά ε, στην μεταρρύθμιση του Ομπάμα για το σύστημα υγείας. Ποιες είναι λοιπόν οι συζητήσεις που γίνονται για αυτό το θέμα. Επίσης, το θέμα της κούρσας των εξοπλισμών ε, μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, το θέμα της Ινδικής ατομικής ε, βόμβας ε, πρόκειται για κάτι το πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Θέλω να ξέρω ποια είναι η συζήτηση που γίνεται στα πλαίσια των πακιστανικών και ινδικών ελίτ πώς αντιδρούν σε αυτήν την ε, διαφορετική ε, θέση και προσέγγιση της ε, Αμερικανικής δίκησης ο πρέσβης. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω τις ερωτήσεις ανά θέμα. Λοιπόν, ερωτήθηκε τι σχέσεις υπάρχουν με, την Ισρα... με το Ισραήλ, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν και τη Ρωσία και ένα ερώτημα για το αν είπα, πρόκειται να επικυρώσουν ή να εγκρίνουν τη συνθήκη αυτή. Και ο κύριος Φόμποντα ρώτησε τι θα μπορούσαν οι ενωσιακές χώρες να κάνουν. Λοιπόν, πρώτον η επικύρωση από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτή επίκειται, αλλά χώρες σαν την Κίνα και την Ινδονησία δεν χρειάζεται να την περιμένουν. Λένε ότι και αυτές θα επικυρώσουν, αλλά περιμένουν την Αμερικανική επικύρωση. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς πολιτικά να πει στις χώρες αυτές να μην περιμένουν την Αμερικανική επικύρωση, ότι δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο. Αυτές όμως περιμένουν. Χρειάζονται 67 ψήφοι υπέρ στην Αμερικανική Γερουσία για την επικύρωση. Και οι δημοκράτες διαθέτουν 65. Κατανοείται βέβαια ότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, είναι και τα υγειονομικά, και οι εσωτερικές ανάγκες της οικονομίας, η κρίση, οι κλιματολογικές αλλαγές κτλ. Και εκεί η Γερουσία πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα μαζί. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να προβλέψουμε τι πλειοψηφία θα προκύψει στη Γερουσία ως προς το θέμα μας και αν κάποιο κόμμα θα ξεπεράσει την κομματική του γραμμή ή όχι. Ο υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός ε, έχει βέβαια με πολλές σχέσεις με τη Γερουσία και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που πρέπει και μπορεί να παίξει αυτή για την επικύρωση και Γενικά μπορούμε να πούμε ότι και τα δύο κόμματα υποστηρίζουν τη συνθήκη. Είτε μπορεί κανείς να την πει δικοματική είτε υπερκομματική. Πρόκειται εδώ για μία στάση κατανόησης της ανάγκης να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα. Όταν αναφέρομαι στον Κίσιγκερ, ο οποίος έλαβε κάποια φιλική προς αυτήν θέση, δεν ε, εννοώ ότι ο Χένρι Κίσιγκερ υποστηρίζει ορισμένους γραφειοκράτες ε, κατά του υπέρ του αφοπλισμού. Όχι. Η στάση τους είναι η εξής. Λένε ότι τα πυρηνικά όπλα είναι τελικά μάλλον αρνητικά στοιχεία στην άμυνα παρά θετικά γιατί μπορεί να υπάρξει εύκολη κατάχρηση τους όχι των ίδιων των όπλων αλλά της τεχνολογίας τους της τεχνολογίας της πυρηνικής σύνδεξης δηλαδή ή του χασίμου υλικού και μπορεί εκεί να τα χρησιμοποιήσουν διάφοροι εγκληματίες. Αν παρακολουθήσατε την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Χένρι Κίσιγκερ και ο Σούλτς παρίσταντο εκεί μαζί με τον Πέρι για να δείξουν ότι πρόκειται για υπερκομματική προσέγγιση. Αυτό ελπίζουμε και εμείς να επηρεαστεί από την υπερκομματική αυτή στάση και η γερουσία στο σύνολό της και να επικυρώσει όπως ζήτησαν ο Σούλτς, Κίσιγκερ και άλλοι. Η συζήτηση στη Γερουσία βέβαια θα εξαρτηθεί όπως είπα και από άλλα θέματα, από τη γενικότερη προσέγγιση της κυβέρνησης για τα πυρηνικά, το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν τα πυρηνικά όπλα στη γενικότερη άμυνα, τον αφοπλισμό κτλ υπάρχει μία μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές μέρες και εγώ ήμουνα στη Washington στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων που λέει ότι θα ήταν θετική η κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια και από επιστήμονες και από πολιτικούς για έγκριση και επικύρωση πρέπει να περιμένουμε χωρίς να υπησέλθουμε στα εσωτερικά των ΙΠΑ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει κάθε χώρα μόνη της να αποφασίσει αν η συνθήκη αυτή τη συμφέρει. Δεν χρειάζεται μια διεθνής γραφειοκρατία ή οργάνωση να την εγκρίνει, αλλά κάθε χώρα. Πρώτα, πρώτα πρέπει να καταλάβει ότι είναι θετικός ο πυρηνικός αφοπλισμός για την άμυνά της, για την ασφάλειά της. Αντί να κοιτάζει κάθε χώρα ποιος άλλος θα την επικυρώσει ή όχι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το έχουν καταλάβει ο Σούλτς και ο Κίσιγκερ. Και πρέπει να το καταλάβει ας πούμε και η Ινδία. μετά τις επιθέσεις στο Μομπάι η Ινδία πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατάχρησης σχασίμου υλικού ας πούμε καθώς και στο Πακιστάν γιατί υπάρχει ανταγωνισμός των εξοπλισμών και μεταξύ των δύο χωρών και φυσικά δεν είναι μόνος τέτοιος ανταγωνισμός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν αλλά και Ινδίας και Κίνας. Πρέπει να γνωρίζει κανείς λοιπόν πόσες εγκατα... πυρηνικές εγκαταστάσεις υπάρχουν, τι όγκος χασίμου υλικού είναι διαθέσιμος και πρέπει ο καθένας να ξέρει τους κινδύνους. Στα πλαίσια λοιπόν των γεγονότων του Μομπάι, για να αποφευχθούν δηλαδή τέτοια είδους γεγονότα στο μέλλον, όπως λέει και ο Σούλτς και ο Κίσιγκερ, πρέπει να καταλάβουν ότι ο μόνος τρόπος είναι να, αποφε... να μειωθούν τα πυρηνικά όπλα για να υπάρχει λιγότερη ή καθόλου δυνατότητα κατάχρησής τους. Είναι βέβαια παλαιό και κλασικό αντικίνητρο αυτό, αλλά είναι αληθινό. δεν είναι καμιά κοινοτοπία. Θυμηθείτε τι έγινε και στο Καρκίλ το 2002 όπου ο Ινδός Υπουργός Αμήνης είπε ότι η Ινδία αν είχε περισσότερα πυρηνικά αύριο δεν θα υπήρχε Πακιστάν. Αυτά δεν τα θέλουμε, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Γιατί υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις στην περιοχή, όχι μόνο πολιτικές και στρατιωτικές αλλά και οικονομικές. Πρέπει λοιπόν η Ινδία, το Πακιστάν, η Κίνα και άλλες χώρες να καταλάβουν τη στάση αυτή και ταυτόχρονα ότι το σημαντικό είναι προς τα που κινείται κάθε χώρα. Η Ινδία πριν απο δυο δυο-τρεις εβδομάδες δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερες δοκιμές βόμβα συντρογόνου. Οι δε Ινδοί επιστήμονες που ήταν υπεύθυνοι για τα πυρηνικές δοκιμές του 1998 το αρνήθηκαν. Είπαν όχι, δεν θέλουμε να βλάψουμε με τις δοκιμές αυτές τις σχέσεις Ινδίας είπα διότι έτσι θα παραβιάσουμε τη συμφωνία 1, 2, 3 είπα Ινδίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι το σχόλιο αυτό δεν προέρχεται από έξω, ούτε από τις Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε από διεθνείς οργανώσεις, αλλά από τους ίδιους τους Ινδούς επιστήμονες. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια ζήμωση, υπάρχουν συζητήσεις. Πολίτες, πολιτικοί και επιστήμονες προσπαθούν να δουν τι γίνεται. Και αυτό είναι μια ένδειξη του τι συμβαίνει γιατί κάτι ανάλογο πρέπει να συμβαίνει και στην Κίνα γίνεται αξιολόγηση των εθνικών συμφερόντων άμυνα ασφαλείας της Ινδίας και εδώ μπορεί πάλι οι πολιτικοί να επηρεάσουν και να είναι χρήσιμοι. Η συνθήκη αυτή λοιπόν μπορεί να εγκριθεί και να τεθεί ενισχύει μόνο αν υπάρξει πολιτική υποστήριξη όχι μόνο από κοινοβουλευτικούς και υπουργούς αλλά και από προέδρους και πρωθυπουργούς. Το 1996 την πρώτη φορά που υπογράφηκε ανάλογη συνθήκη δεν είχε χρειαστεί η υποστήριξη του Κλίντον, του Σιράκ ή του Μέιτζορ γιατί εκείνοι γνώριζαν ότι ήταν απαραίτητη και σε λιγότερο από τρία χρόνια από το μηδέν επικυρώθηκε η συνθήκη αυτή και γιατί όχι γιατί οι πρεσβευτές σαν και εμένα έπεισαν τους πολιτικούς αλλά γιατί η ίδια η πολιτική ηγεσία ήταν πεπισμένη τέτοιου είδους λοιπόν δέσμευση χρειάζεται αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων Κάποιος μίλησε τώρα για το Ισραήλ. Το Ισραήλ σε υπουργική διάσκεψη που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με 40 υπουργούς και τη Χίλαρη Κλίντον και άλλους το Ισραήλ δήλωσε ότι ε, δεν είπε μεν ρητά ναι ότι θα επικυρώσει τη συνθήκη αν και την έχει υπογράψει αλλά είπε ότι αν το σύστημα είναι λίγο πυκνότερο, τότε θα μπορούσαμε να επικυρώσουμε και κάτι με δεν είναι δύσκολο να γίνουν οι αλλαγές που ζητάει το Ισραήλ. Άρα είναι δυνατόν να συνδυαστούν οι προσδοκίες με την επικείμενη επικύρωση από τη ΣΥΠΑ. Και υπάρχει μεγάλη πίεση προς το Ισραήλ να επικυρώσει Στα πλαίσια βέβαια της γνωστής σύραξης και διαφορά στη Μέση Ανατολή υπάρχει και η στήριξη των αδεσμεύτων Για τη Ρωσία, η Ρωσία επικύρωσε τη συνθήκη, δεν προέβλεψε τόσους πολλούς σταθμούς όσο η ΕΠΑ, 90% ζήτησε η Ρωσία, η 60% μόνο η Ρωσία, και αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει υπόδειγμα, παράδειγμα και για την Κίνα. Αν η Ρωσία λοιπόν επικυρώσει επίσημα πριν από τη ΣΥΠΑ, αυτό θα ενθαρρύνει και την Κίνα. Ο ρόλος των πυρηνικών όπλων τώρα Δεν θέλω να σας επιβάλλω τη δική μου άποψη και κρίση. Αναφέρομαι στα λόγια του ε, Χένερι Κίσιγκερ για πλήρη κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Αν θα, η συνθήκη αυτή θα το πετύχει είναι αμφίβολο, αλλά μετά τη συνθήκη Start, μετά τις περικοπές που έγινε και το σύστημα επαλήθευσης θα πρέπει να λυθούν ορισμένα δευτερεύοντα υποστρατηγικά θέματα και το πυρηνικό πλωστάσιο όλων των χωρών τουλάχιστον να μειωθεί. Είναι ένα βήμα δηλαδή. Ένας συνδυασμός όλων αυτών που θα μας οδηγήσει προοδευτικά, μπορεί να μας οδηγήσει προοδευτικά προς τον πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό. Υπάρχει κίνηση πάντως και συζήτηση των ιδεών αυτών. Τέλη Δεκεμβρίου θα ξανασυζητηθεί η νέα συνθήκη START και το σημαντικό είναι να μην μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Βέβαια ε, η προσωπική μου άποψη δεν είναι ίσως οικουμενική αλλά φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε πάρει τη συνήθεια να περιμένουμε τους άλλους. Η δήλωση του Ομπάμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν ότι μας κατηγορήσατε όλοι ότι δεν συζητούμε το θέμα, τώρα που το συζητούμε πρέπει και εσείς να μας υποστηρίξετε. Επρόκειτο δηλαδή για έκκληση, για κοινή δράση, γιατί όντως είναι ευθύνη όλων μας να βοηθήσουμε ενεργά σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, ένας από τους οποίους είναι ακριβώς η επικύρωση της συνθήκης αυτής όχι στις ε, πρωτεύουσες της Ένωσης, γιατί η Ένωση θα επικυρώσει, αλλά περίπου όπως είπε ο κύριος Σιβόμποντα. Εμείς συνεργαζόμαστε με κοινοβουλευτικούς, με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση, με εμπειρογνώμονες και ομιλητές. Υπάρχει πολύ μεγάλη δικτύωση. Και εσείς μπορείτε έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε μέσω του δικτύου και του διαδικτύου με ανθρώπους στον Τάρε Σαλάμ, στην Ινδονησία και αλλού. Σε κάθε χώρα όπου γίνεται προσπάθεια επικύρωσης. Τέτοιου είδους πράγματα μπορείτε να κάνετε και μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πιο ενεργοί. Άλλος ρώτησε για ο κύριος Γκαλτιέρη μίλησε για ελπίδα και απελπισία. Το hope, η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η καταιγίδα των τελευταίων δέκα ετών οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι θετικές. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να προχωρήσουμε και δεν χρειάζεται αναβίωση της συνθήκης αυτής γιατί αν και οι 150 επικυρώσεις της δείχνουν ότι η οργάνωση είναι ακόμη ζωντανή. Χρειάζονται μόνο τα τελευταία βήματα. Θα μπορούσα να σας δείξω δύο-τρεις διαφάνειες αν χρειάζεται. Αν δείτε σε ποιους τομείς ε, εμφανίζεται η πυρηνική τεχνολογία θα διαπιστώσετε ότι στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική κυρίως υπάρχει εξέλιξη των πυρηνικών. Και αν σε αυτόν το χάρτη, αυτόν το χάρτη τον συγκρίνεται με τις περιφέρειες, περιοχές όπου γίνεται προσπάθεια μείωσης των πυρηνικών, θα δείτε ότι εκεί που λείπει τέτοια υποστήριξη είναι στην Ασία, τη Μέση Ανατολή επίσης και τη Λατινική Αμερική. Άρα Εκεί ακριβώς λείπουν και οι περισσότερες επικυρώσεις στην Ασία και τη Μέση Ανατολία. Πράγμα που μας θυμίζει ότι δεν θέλει κανείς να υπάρξει το λεγόμενο πυρηνικό μποτιλιάρισμα bottleneck γιατί αν η πυρηνική ενέργεια αναπτύσσεται κατά 12% το χρόνο στην Ασία και 10% στη Μέση Ανατολή, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας θα ανταποκρίνονται σε αυτού του είδους τα γεγονότα. Ότι θα ζητάμε δηλαδή και την ανάλογη μείωση. Να, εδώ, εδώ βλέπετε τις διαφάνειες. και από εκεί φαίνεται πού μπορεί να χρειάζεται περισσότερη επαλήθευση και επιτήρηση. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Λέτε αυτό το οποίο υπογράμμισε και ο συνάδελφος Σβόμποντα. Ε, αν τα κράτη-μέλη δεν επικυρώσουν αυτήν την ε, συνθήκη για τα μάτια ενός πρέσβη, καταλαβαίνετε ότι δεν θα την επικυρώσουν ούτε και για τα μάτια των Ευρωβουλευτών. Μέσα από τα διάφορα δίκτυα και τις εργασίες των διαφόρων διακοινοβουλευτικών επιτροπών πρέπει να προωθήσουμε όλη αυτή την ε, λογική και να το παλέψουμε. Η κυρία Νικολάη. Κύριε Πρέσβη, δεν μπορώ να αγνοήσω ότι για αυτήν τη συνθήκη ε, ε, εξαντλήσαμε πολύ διπλωματία ε, και ασκήσαμε και πολύ πίεση, ψυχολογική πίεση. Αλλά ακόμη κι αν η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε την επικυρώσουν, παραμένει πάντοτε ο έλεγχος αυτών των χωρών, μάλλον των χωρών εκείνων που θέλουν να μπλοκάρουν την συνθήκη αυτή. Υπάρχει αυτή η φόρμουλα τη συνθήκη στο άρθρο 14 που μπλοκάρει πραγματικά την εφαρμογή. Εσείς πιστεύετε ότι η τροποποίηση αυτού του άρθρου θα μπορούσε να βοηθήσει η κυρία Λούνετσεκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε παρόν εδώ κύριε Πρέσβη και λυπούμε που, και ζητώ συγγνώμη που δεν παριστάμουν ε, στην αρχή της ομιλίας σας αλλά ε, είμαι νεοεκλεγής Ευρωβουλευτήνα αλλά σαν, ε, σαν βουλευτήνα στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Αυστρίας σας παρακολουθούσα. Έχω δηλαδή μια ιδέα περί του τι κάνετε. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο πράγματα εν ονόματι των Πρασίνων και της ομάδος Αυτά τα οποία λέτε όντως μας εξηγούν τι γίνεται. Δηλαδή, αν ο καιρός είναι καλός, μπορεί κανείς να πάει στη διοπλοεία. Λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να υποφεληθεί από το ότι έχει κάνει ο Ομπάμα τελευταίος για να έχουμε αποτελέσματα και να λειτουργήσει αυτό, αυτή η συνθήκη. Σχετικά με αυτό που ρώτησε πριν ο κύριος Λόμποντα και εγώ πιστεύω ότι σαν βουλευτές στις συνεδριάσεις μας μπορούμε στις συναντήσεις που έχουμε με οι κοινοβουλευτικούς από διάφορες χώρες να υπογράψουμε ότι υπάρχει ανάγκη να κυρωθεί η συνθήκη αυτές προς όφελος των ε, χωρών που ενδεχομένως δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν έχω πλέον ερωτήσεις, ήθελα απλούστατα να σας πω ότι σας υποστηρίζω πλήρως και εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτά τα οποία ε, είπατε. Ευχαριστώ. Σχετικά με το, τον τύπο ε, που θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή ε, είναι κάτι που έχει καθοριστεί και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως σας είπα υπάρχουν 44 ονόματα και χρειάζονται όλες οι κυρώσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Καταρχήν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι τελείως απρόβλεπτοι όπως ξέρετε και ε, πεισματάριδες οπότε δεν θα είναι εύκολο να διαβλέψουμε τώρα ε, πότε θα ε, υπάρξει κύρωση. Το ερώτημα είναι πρέπει η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα να είναι όμοιρος αυτής της συνθήκης. Εγώ θα μπορούσα να το αντιστρέψω και να πω ε, εάν ε, ελέγξουμε αυτή τη συνθήκη βλέπουμε ότι βελτιώνεται με κάθε δοκιμή ε, διότι βοηθάει στο να δημιουργούν μικρότερες μικρότερους εξοπλισμούς για να κάνουν τις δοκιμές και η τεχνολογία η οποία προφανώς ενδιαφέρει και ανησυχεί τις χώρες της περιοχής με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διαδίδεται ε, είναι κάτι που μπορεί να με υπενθυμίσει σε όλους μας ότι δεν μιλάμε μόνο για το δυνητικό πρόγραμμα επέκτασης το οποίο θα επηρεάσει μόνο χώρες μιας συγκεκριμένης περιοχής αλλά ε, αν ε, αν γίνει ένα ξεπούλημα προς κάθε ενδιαφερόμενο είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί όλους μας διότι ενδεχομένως ε, αυτοί οι οποίοι θα μείνουν πίσω ε, θα ε, υπονομεύσουν το οικοδόμημα. Μία χώρα λοιπόν μπορεί να κάνει μία δοκιμή στο χωράφι κάποιου άλλου θα μπορούσε ίσως ε, να ε, να υπάρξει υπεργολαβία και πώληση υπηρεσιών προς άλλους και ε, αντί να σκεφτόμαστε ότι χρειαζόμαστε 7 ε, κυρώσεις ακόμη θα χρειαστεί ε, να γίνει μια επιπρόσθετη προσπάθεια. Ίσως είναι αφελές αλλά αν δεν ήταν ε, αφελές το 1996 να διαβλέψει κανείς την κύρωση αυτής της συνθήκης δεν νομίζω ότι είναι πλέον ανόητο να σκεφτούμε ότι δεν μπορεί να κυρωθεί. Βέβαια χρειάζεται ε, ε, ενέργειες, χρειάζεται την παρουσία πολιτικών ηγετών αλλά προσπαθώ να σας προσιλητήσω εάν μου επιτρέπετε θετικά βέβαια ε, και να σας πω ότι είναι κάτι που δεν αναφέρεται σε εμά, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς αυτό είπα και στους συναδέλφους στη Γενέβη πίσω από κάθε βήμα που κάνουμε ε, υπάρχει, υπάρχει ένας λόγος και θα πρέπει να μπορέσουμε ε, να προχωρήσουμε ε, μόνο με θετική συμμετοχή. Όχι να βραχικυκλώσουμε το σύστημα. Ε, το σύστημα αυτό λειτουργεί ε, και ίσως θεωρήστε ότι δεν είναι ανάγκη να ισχύσει η συνθήκη αλλά δεν νομίζω ότι είναι θετική αντιμετώπιση διότι πρέπει να αντιληφθούμε και δεν θέλω να το επαναλαμβάνω συνέχεια ότι δεν είναι ευκαιρία για διμερείς αντιμετωπίσεις. Αυτό που είπε και δεν είπε ο κύριος Ομπάμα ήταν παρακαλώ όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τρία χρόνια ίσως ε, και σε λιγότερο χρονικό διάστημα ε, στις εκλογές σε δυόμιση χρόνια η Αμερική η ε, Αμερικανοί πολιτικοί να πιεστούν να, από τους πολίτες για τα ωφέλη για τις δυνατότητες του συστήματος και να πιεστούν. Ε, βέβαια η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 1996. Άρα πρέπει να δείξει κανείς συγκεκριμένα ότι υπάρχει μία επένδυση η οποία αποδίδει. Διαφορετικά θα χρειαστούν δεκαετίες μέχρι ότου επανέλθει ο, ο ήλιος και αντιληφθούμε ότι η ιστιοπλοεία καλύτερα εξασκείται στη Λιακάδα από ότι στη Θεομηνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρέσβη. Αυτή η διδακτική συνεδρίαση ήταν πολύτιμη για όλους. θα σας ακούσουμε και σε άλλες φάσεις όλου αυτού του σχεδίου όπου το Κοινοβούλιο θα παίξει σημαντικό ρόλο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στενή επαφή και σας καλώ να ξανάρθετε του χρόνου για να μας πληροφορήσετε και πάλι για αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε στις 15 Οκτωβρίου και θα ακούσουμε τον κύριο Βάης από την ε, Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αφοπλισμού και στις 6 Οκτωβρίου θα ακούσουμε τον κύριο Σέκη, τον ε, απεσταλμένο στο Αφγανιστάν. Παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν για λίγο. Θα συνεχίσουμε την ε, συνεδρίαση που αφήσαμε ανοιχτή χθες.